της έχω λάβει ε, προτάσεις από το Συμβούλιο για τις ε, προτάσεις της Επιτροπής που επίσης έχουν διανεμηθεί και θα διανεμηθούν στο Κοινοβούλιο. Η περίοδος για την κατάθεση των προτάσεων αρχίζει αύριο. Και στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής της διάταξης που είναι τα ζητήματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκινάμε με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη. Δίνω το λόγο πρώτα στους συντάκτες των, του ψηφίσματος. Κυρία Ντεκεζέχ, καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ταϊλάνδη